Έχω βέβαια κάποιες ανακοινώσεις να σας κάνω στα τσεχικά, λέει ο Πρόεδρος. Έχω λάβει τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την πρώτη ανάγνωση και τις ε, αιτιολογήσεις ε, επίσης, τα ονόματα θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά. Η περίοδος των τριών μηνών θα ξεκινήσει από αύριο, 30 Σεπτεμβρίου δηλαδή 2011. Thanks a lot. Now we will continue with the... Συνεχίζουμε τώρα με τις επεξηγήσεις